Λοιπόν, κηρύσω την έναρξη σημερινή μα συνεδρίαση. Έχουμε 10 λεπτά καθυστέρηση, διότι ανάμεσα στη συνεδρίαση των συντονιστών και τη συνεδρίαση της Επιτροπή μα τη δημόσια, έπρεπε να βάλει μπρο το σύστημα webstream για να μεταδιδόμαστε και στο διαδίκτυο. Και ε, σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Σας καλωσορίζω. Είναι σύντομη σχετικά η ημερήσια διάταξη σήμερα, αρκετά βραχία. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτα επιθυμίε για αλλαγή τη ημερήσια διάταξη. Ποιος θέλει. Όχι, τίποτα, τίποτα. Καλώ. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ανακοινώσει του Προέδρου. Σύντομα θέλω να σας πω ότι αποφασίσαμε στη συνεδρία των συντονιστών τα εξής. Επειδή χτες οι διαπραγματεύσεις για τους συμβιβασμούς ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με μεγάλη επιτυχία. Ε, διατηρούμε την ε, ψηφοφορία για την Τετάρτη, την ερχόμενη. Αν δεν υπάρξουν μεγάλα προβλήματα μέχρι την Τρίτη που είναι η τελευταία τεχνική συνεδρίαση, σε περίπτωση που προκύψει κανένα πρόβλημα, θα αποφασίσουμε την άλλη εβδομάδα πότε θα αποφασίσουμε. 8 Δεκεμβρίου λίγη εντολή μας και μέχρι τότε θα πρέπει να καταθέσουμε την τελική έκθεση και η τελική ψηφοφορία της έκθεσης με τις συστάσεις των πολιτικών ομάδων προβλέπεται για την Σύνοδο Ολομελίας του Δεκεμβρίου. Έχουμε κάποιο περιθώριο χρονικό. Αυτό ήταν το πρώτο. Την άλλη εβδομάδα ψηφίζουμε. Δεύτερο, η γραμματεία δεσμεύτηκε να στείλει σε όλους τους καταλόγους ψηφοφορίας και τις συμβαστικές τροπολογίες ε, ακόμα τούτη τη βδομάδα για να μπορέσετε όλοι να προετοιμαστείτε γιατί είναι πολλές οι τροπολογίες και οι προσωπικές επιθυμίες γενικότερα που εκφράζονται. Και μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα μπορείτε να το συζητήσετε και με τις ομάδες σας και να το σκεφτείτε. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αποφασίσαμε στην τρίτη την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου να κάνουμε άλλη μια ακρόαση και μια τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών. Η επιπλέον ακρόαση έχει στόχο να ξανασυζητήσουμε δημόσια το, το θέμα του Αζερβαϊτζάν, το Λανδρομάτ και τη Σλοβενία, όπου το, Σλοβενικό Κοινοβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αρχίσουν ε, έρευνες ε, των διοκτικών αρχών ε, για νομοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες, κοινό ξέπλυμα. Κάποια άλλα θέματα μάθαμε χθε για την Πορτογαλία ότι ξεκίνησαν διώξει για πρώην υπουργού σε σχέση με τα έγγραφα του Πάναμα. Αυτό δεν θα φτάσει στην ακρόαση τη δική μα, επειδή εμεί εξαρτώμαστε από τι δημοσιεύσει του δικτύου των δημοσιογράφων. Θα ε, μας φαίνουν περιπτώσεις και στο μέλλον, περιπτώσεις για τις οποίες εμείς δεν έχουμε πρόσβαση όμως στα αυθεντικά έγγραφα. Και... Τελικά στην Ολομέλεια Ε, είναι στα χέρια των πολιτικών ομάδων τι θα παρουσιάσουμε μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης. Έχουμε χρόνο μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου να συζητήσουν οι πολιτικές ομάδες ε, τι ε, συνέχεια θέλουμε να δώσουμε για την ομοθεσία φυσικά. Αυτά είναι θέματα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και ΕΚΟΝ. Για τη διοργανική συμφωνία αυτά είναι στα χέρια των πολιτικών ομάδων και από εκεί και πέρα για άλλα συμπεράσματα και δράσεις, ας πούμε, ίδρυση η σύσταση νέων επιτροπών, ε, εξεταστικών επιτροπών, αρμοδιοτήτων των επιτροπών και πάλι αυτά είναι στα χέρια της Ολομέλειας πια. Αυτά τα συμπεράσματα θα προετοιμαστούν ε, από τις πολιτικές ομάδες. Τελευταίο. Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση που θα κάθεται εδώ ο Αντιπρόεδρος Φάμπιο Ντεμάζη και γενικά στο Κοινοβούλιο. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την ενεργή ε, παρουσία του. Δεν συμφωνούσαμε πάντα 100%. Ήταν όμως επικοδημητική η στάση του. Ε, του εύχομαι καλή επιτυχία ε, στη Γερμανία, στην Bundestag ω μέλο τη Γερμανικής Βουλής πλέον από τα νέα του καθήκοντα. Και πάμε τώρα στην ημερήσια διάταξή μας στο σημείο 3 που θα συζητήσουμε τις τροπολογίες που έχουμε για τις δύο εκθέσεις. Θα δώσω το λόγο στο Γέπε Κόφωτ. Thank you so much, Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους των εισηγητών, δεν μπορούσε να αναδώ μέρος ο συνάδελφος, σας ευχαριστώ όλου για, για τις τόσες πολλές τοπολογίες, τα 350 για τα ευρήματά μας και τις συστάσεις μας, για την έκθεσή μας. Τις εξετάσαμε προσεκτικά. Πολλέ είναι πολύ καλές και έχουν βελτιώσει τη δουλειά μας ως εισηγητών. Να ευχαριστήσω και τους Κιώδη για την πολύ ενεργό συμμετοχή τους στην σύνταξη. και για να βρούμε συμβιβαστικέ λύσει. Είχαμε πολλέ ε, συζητήσει των σκιωδών εισηγητών, πολλέ συναντήσει. Χθε μόλι συναντηθήκαμε για πάνω από τρει ώρε και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την πολιτική μα δουλειά. Τώρα λοιπόν έχουμε συμβαστικέ τροπολογίε για τα βασικότερα πολιτικά ζητήματα στην εκθεσή μα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων ω εδώ. Δεν θα μπω σε όλε τι λεπτομέρειε, απλώ θα πω ότι είναι σαφές για όλους μας, ε, ιδίω για μένα ως εισηγητή, ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά μας εδώ για την νομιμοποίηση των παράνομων προσόδων, για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ε, και καλώς ε, αναφέραμε στην αρχή της συνεδρίασης ότι διαρκώς προκύπτουν νέες υποθέσεις καθημερινά. Παρόλο λοιπόν που έχουμε κάνει τεράστια δουλειά σε αυτή την Επιτροπή, με τι ακροάσει μα, τι αποστολέ μα, ε, την δουλειά μα εδώ, για μένα είναι πέρα αμφιβολία ότι η εξακολούθηση του θέματο, ε, τη προσοχή μα επί του θέματο, είναι σημαντική ε, για να ασκούμε διαρκώ πίεση για να αποφεύγουμε την νομιμοποίηση παράνομων προσόδων, την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Θα συζητηθεί έκθεση το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια, αλλά είναι ένα θέμα τόσο σημαντικό γιατί ήδη δείχνει την αξία το έργο, του, το έργο που κάναμε. Ήδη υπάρχουν αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από άλλου και πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Απλώ να ακούσω προσεκτικά του συναδέλφου τη Επιτροπή, τα δικά του σχόλια και πραγματικά ανυπομονούμε για την περαιτέρω συνεργασία μα και σε αυτή την Επιτροπή και ελπίζουμε και σε έναν ε, μελλοντικό ε, σχηματισμό στο μέλλον. Ευχαριστώ. απουσιάζει σήμερα. Νομίζω για θέματα εσωτερικής πολιτικής είναι στην Τσεχική Δημοκρατία. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Έχω άλλη μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους. Στην επεξεργασία των συμβαστικών προτάσεων και τροπολογιών, καλύψαμε όλες τις συστάσεις. Για όλες τις συστάσεις υπάρχει ένα συμβιβασμό. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, όταν τελειώσει η ψηφοφορία και και εγκρίνουμε τις συμβαστικές προτάσεις, θα έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφορίας υποφερτό, εν πάση Οι τροπολογίες ήταν πάνω από 1.400, 667 συν 783. Μπορείς να πεις τίποτα γι' αυτό, σε παρακαλώ, Γεπέ, ως εισηγητής. Yeah, it, ναι. Στις συμβαστικές κοιτάξαμε να καλύψουμε όλα τα εδάφια. Κάποιες είναι πιο σημαντικές. Σε κάποια σημεία παραμείναμε στο αρχικό κείμενο, αλλά μόνο αφού υπήρξε συμφωνία μετα... μεταξύ των σκιωδών. Σημαντικό να υπογραμμιστεί και αυτό. Ουσιαστικά ε, όλα τα εδάφια ε, έχουν ε, μια συμβαστική που τους αντιστοιχεί και λάβαμε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Την απάτη καταπολεμάμε εδώ. Και να τονίσω ότι για μα είναι σημαντικό ότι είναι έκθεση εξεταστική επιτροπή. Δεν είναι μια παραδοσιακή έκθεση επιτροπή. Είναι ειδική έκθεση, οπότε κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ευρεία συνένεση και μα υποστηρίζουν όλοι. Ε, τα ευρήματα τη επιτροπή είναι σημαντικά. Οπότε είναι σημαντικό τα ευρήματα αυτά να διατυπωθούν με τρόπο να καλυφθούν όλα τα έγγραφα που ανακαλύψαμε, να αντικατοπτρίζουν αυτό στις συστάσεις μας. Πρόεδρε, θα μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες για τις τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι θα μας έπαιρνε όλη τη συνεδρίαση, αν τις αναλύσω. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει καλές συμβαστικές λύσεις για τα βασικά ζητήματα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης ηγητές τώρα. Πρώτος ο κύριος Νίτερ, Μάγερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω όχι μόνο τους εισηγητές, αλλά και την τεράστια δουλειά του προσωπικού των πολιτικών ομάδων και της γραμματείας. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο γενικότερα Νομίζω ότι το θέμα αυτό αφορά, είναι μία από τις μεγάλες ε, προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία, για την ε, ε, φορολογική κατάσταση, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση αδικίας, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σημαντικό, γιατί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ένα ρόλο στη βελτίωση της κατάστασης σε όλο τον κόσμο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πολύ περήφανο για τη δουλειά του στον τομέα αυτό κατά τα τελευταία χρόνια. Τα έγγραφα του Παναμά είναι λίγο διαφορετικά από το LuxLeaks. Είναι ε, διαφορετικά καλύπτουν μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο κατά την οποία υπήρξαν ε, ουσιαστικές αλλαγές νομοθεσίας ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλύπτουν επίσης ε, πολύ ευρύτερα ζητήματα και συνεπώς αυτά που μαθαίνουμε είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μη ευρωπαϊκών εταιριών που φαίνεται να προωθούν πρακτικές οποίες εμείς θεωρούμε εσφαλμένες και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις ε, μεταφορά χρημάτων στις εταιρείες όπως μάθαμε για παράδειγμα από τις διαρροές για τα έγγραφα του Παναμά, μάθαμε να ενδεχομένως να ε, είναι και υπό τις ευλογίες ε, των κυβερνήσεων των χωρών. Επιτρέπεται δηλαδή ασφαλής πρόσβαση ε, στον, στα χρήματα αυτά, τα οποία μένουν στο περιθώριο της νόμιμης οικονομίας. Λοιπόν, σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή μας νομίζω ότι έχει συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες, έχει αποκτήσει βαθιά γνώση ε, για την κατάσταση και νομίζω ότι μπορούμε να την αξιοποιήσουμε όχι μόνο εμείς ως Ευρωβουλευτές, αλλά και οι πολίτες μας και ολόκληρη η κοινωνία. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά φιλόδοξο, όπως συχνά λέμε στο Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο στόχος είναι κοινός από τη έχω καταλάβει από τις ε, συνεδριάσεις των σκιωδών. Θέλω να έχουμε μια καλή έκθεση η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έμπνευση και που θα μπορέσει να τύχει μεγάλη υποστήριξης. Και όπως είπε και ο εισηγητής, υπήρξε πολιτική συμφωνία, αλλά η διατύπωση σε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες ε, παραμένει εκκρεμής. Από ό,τι κατάλαβα βέβαια, αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι κατά τις ε, συναντήσεις συμφωνούμε ε, με την πρόκληση υπάρχει μια ε, κοινή, ε, υπάρχει μια υποστήριξη, να υπάρξει μια κοινή διατύπωση που θα μπορεί να υποστηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Να υπάρξει δηλαδή ένα συμβιβασμός που θα, είναι, που θα προτείνει εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις. Να τονίσω μερικά σημεία τα οποία θεωρώ αρκετά σημαντικά. Πρώτον, Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των αθέμητων πρακτικών και των ε, πρακτικών μερικές φορές ε, δυστυχώς ε, είναι νόμιμες γιατί είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση για το παράνομο πρέπει να υπάρχει καλύτερη επιβολή του νόμου ε, ενώ στην άλλη περίπτωση πρέπει να δούμε κατά πόσο ο σχεδιασμός της νομοθεσίας είναι καλός και υπάρχει περισσότερο, μεγαλύτερο περιθώριο βελτιώσεων. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει νέα νομοθεσία ή νέοι φορείς, να δούμε τι έχουμε στη διάθεσή μας και να δούμε κατά πόσο λειτουργούν σωστά και όπως πρέπει. Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχουν παραθυράκια ε, τα οποία θα αφήσουμε ακάλυπτα. Εγώ νομίζω ότι ο κώδικας ε, δεοντολογίας ε, που θέλουμε να προωθήσουμε όντως πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να ζητήσουμε τη βελτίωσή του. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την ε, πορεία της όλης, να σχεδιάσουμε την πορεία της όλης διαδικασίας. Είναι όμως πολύ καλό σημείο αφετηρίας για τη δουλειά μας και πρέπει απλώς να το, τη βελτιώσουμε, να υπάρξει μια έκθεση που πραγματικά να αξίζει τον κόπο και που θα τύχει υποστήριξη ευρεία μεταξύ των ε, ευρωβουλευτών οι εισηγητές, ε, οι εμπειρογνώμονες και η γραμματεία έκαναν ό,τι μπορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να το πω αυτό. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι να ε, συμβάλλω στην έκθεση της Επιτροπής και ελπίζω επίσης και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε γέρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νίτερμαγερ, ένα σημείο θέλω να υπογραμμίσω και να τονίσω χωρίς να σχολιάζω τα πάντα. Η διάκριση που λέτε μεταξύ φοροαποφυγής και ε, δημιουργικής φορολογικής ε, πολιτικής. Η φοροαποφυγή είναι παράνομη και η φοροδιαφυγή. Ε, τώρα το να έχει μια δημιουργική φορολογική ε, πολιτική ω εταιρεία είναι νόμιμο, αλλά καλή σαν λέξη νομοθεσία. Σοσιαλδημοκράτες, η κυρία Ρέγνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευθύ εξ αρχή ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του δύο εισηγητέ που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, αλλά και όλη την ομάδα και τους κοιόδης εισηγητές ε, που συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης. Θα ήθελα τρία πράγματα να πω έχω πάρα πολλά, αλλά τρία να τονίσω, ε, που μάθαμε εδώ στην Επιτροπή μας για τα έγγραφα του Παναμά. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε ε, τα πιο ε, αμφίβολα σχήματα ε, φοροδιαφυγής και φοροφυγής, να τα γνωρίσουμε και να τα ανακαλύψουμε με διάφορους τρόπους. Δεύτερον, χωρίς τη βοήθεια ιδιωτικών τραπεζών, ορκωτών λογιστών, δικηγόρων κτλ. δεν θα είχαμε τέτοια διαφυγή κεφαλαίων και στο βαθμό που την έχουν. Και τρίτον, δεν θα πρέπει να ενισχυθεί επιγόντως ε, και να αυστηροποιηθεί ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά να ελέγχεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο αυστηρά η κείμενη νομοθεσία. 172 τροπολογίε έχουμε κάνει εμεί οι σοσιαλδημοκράτε για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το σχέδιο έκθεση και γι' αυτό για να επανέλθω στις εταιρείε θηρίδες, μαϊμού. Εκεί υπάρχουν διάφορα κατασκευάσματα και τεχνάσματα, πάρα πολλοί χώρος για δουλειά και ζητάμε και από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να κοιτάξει τι θα γίνει με την νομοθεσία και με το δίκαιο το εταιρικό. Όχι ε, μόνο να μιλάμε για το αγγλοσαξονικό χώρο. Επίσης, τι είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες οι ε, πολυεθνικές χώρο ε, διαφεύγουν και σήμερα και στο μέλλον και αυτό έχουν άμεση σχέση με τη δική μας ε, επιτροπή και σωστά βγήκε στην έκθεση. Και τέλος, η μαύρη λίστα των φορολογικών, όχι παραδείσων, βαλτοτόπων. αλλά έχουμε βρει τέτοια μέρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πρόκειται για τρίτες χώρες είμαστε πολύ γενναιόδοροι και μεγαλόψυχοι και τους ε, έχουμε δακτυλοδεικτούμενους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείτε τι γίνεται. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά. Θα πρέπει επιγόντω όμως να καθαρίσουμε τα το οίκου μα για να μείνουμε και αξιόπιστοι. Και τέλο για τη φορολογική δικαιοσύνη. Σας παραπέμπω στον κύριο Γιούνκερ ε, για την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εκεί υπάρχει πεδίο δράσης. Να πω στους συντηρητικούς συναδέλφους. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ που χάνουμε και μας λείπουν επιγόντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να είναι το κίνητρο, ε, η κινητήρια δύναμη να προχωρούμε ξεκάθαρα και να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, να μην τα λέμε συγκαλυμμένα στην τελική μας έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτά τα χρήματα τα χρειαζόμαστε και μας λείπουν. Δεν είναι 12 παρα 5 εδώ, είναι 12 και 10 αυτό δεν θα πρέπει απλώς να μας ταρακουνήσει, να φυπνιστούμε, αλλά να έχει και αποτελέσματα, έτσι ώστε η δίκαιη φορολογία να μην είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εμάς εδώ φιλολογικά, αλλά να έχει και αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέγνερ. Υπογραμμίζω και είναι υπογράφω όλα αυτά που λέτε. Γιατί το λέτε αυτό στο ΕΛΚ που μας απακολείται και μάλιστα πάντα συντηρητικούς, ε, παραδοσιακά. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχουμε διαφορές. Γιατί προσπαθείτε τεχνητά να δημιουργήσετε διαφορές μεταξύ μας. Ε, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Ο συνάδελφος Τζαμπάσκι εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο. Κυρία Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, το προσωπικό και όλους όσους συμμετείχαν ε, και που ακόμη είναι ενεργοί στην διαδικασία αυτή της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό το πνεύμα, υπήρχε πνεύμα συνεργασίας, φτάσαμε επιτέλους σε αυτό το στάδιο. Τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας εργασίας και όχι το τέλος ε, απλώς μιας ε, διαδικασίας. Θα ήθελα να πω ότι με 700 τροπολογίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψω όλα όσα θα ήθελα να πω. Ε, κάπως επιφανειακά θα τα πω. Υπάρχουν μικρότερη σημασία τροπολογίες ε, διατύπωσης καθαρά και άλλες πιο σημαντικές. Πολλές τροπολογίες όμως ε, περί διατύπωσης βοηθούν Υπάρχουν πολλά, πολλές καλές τροπολογίες ε, για ε, τη Μόσακ Φονσέκα, για τους ε, διαμεσολαβητές και για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων της Ένωσης και των κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεσή μας θα αποτελέσει βάση σημείο αναφοράς και στο μέλλον. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακριβείς και πολύ διεξοδικοί και για αυτό το θέμα αλλά και για άλλα ζητήματα ακόμη και αν αυτό καταλήξει σε μία μακροσκελέστερη έκθεση για τις νέες ε, πρωτοβουλίες ε, που αναφέρονται στις τροπολογίες, σημειώνω με χαρά ότι υπήρχαν πολλές τροπολογίες που τόνισαν τη σημασία ευθυγράμμισης ε, των και των εμπορικών πολιτικών δεν έχουν γίνει αρκετά νομίζω σε αυτό το τομέα ε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πώς γίνεται ο φορολογικός σχεδιασμός και πώς συνδέεται αυτό με την εταιρική ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το City πρέπει να το προσέξουμε όλο ιδιαίτερο, επειδή είναι φορολογικό παράδεισο και είναι σημαντικό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ε, για το Brexit. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Επίση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα ε, σαφή χάρτη πορεία για το πώ θα συνεχίσει η δουλειά τη Επιτροπή Πάνα και πώ θα είναι πιο μόνιμη. Υπήρχαν πολλέ καλέ προτάσει και από αυτό. Κάτι ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πράγματα τα οποία δεν θεωρούσαμε ρεαλιστικά ε, παρόλα αυτά μπορούν να δημορφώσουν ήδη μία βάση για το τι είναι πολιτικό εφικτό όλο αυτό, αυτή η διαφάνεια υπέρ της, η, η, το θεματολόγιο υπέρ της διαφάνειας και κατά των φορολογικών παραδείσων θεωρούσαμε ότι δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν. Ένα ζήτημα που πρέπει να καλύψουμε στο μέλλον είναι ο προβληματικός ρο, ε, ρόλος των τεσσάρων μεγάλων ε, ε, εταιριών ελέγχου γιατί είναι και φορολογικοί σύμβουλοι και ελεγκτές. Ε, και έχουν και άλλους ρόλους. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει. Είναι λοιπόν ε, η έκθεσή μας νομίζω ε, μια πολύ καλή βάση και ελπίζω ότι όλες αυτές οι τροπολογίες θα, θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση. Οι 23 τροπολογίες έχω αφήσει για να τις συζητήσω με τους συναδέλφους, αφορούσαν πολλά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά ε, για παράδειγμα κάποια αποσαφηνίζουν το κείμενο της έκθεσης αλλά συμπεριλαμβάνουν και νέες ε, πρωτοβουλίες ε, που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό να προχωρήσει η θεματολογία της Επιτροπής μας. Κάποια από τα ζητήματα που συζήτησα και με τους συναδέλφους ιδιαίτερος πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει φοροδιαφυγή, τι σημαίνει φοροαποφυγή, τι σημαίνει φορολογική απάτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει απαρκή νομοθεσία για ε, να ε, προστατεύσει τους ε, διερευνητικούς δημοσιογράφους ή τους καταγγέλλοντες των ατασταλιών. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να τονίσουμε επίση το γεγονό, όπω έκανα εγώ με του συναδέλφου, πρέπει οι φορολογικέ και εμπορικέ πολιτικέ ε, να ευθυγραμμιστούν. Ε, νομίζω ότι είναι γνωστό πια ε, η σχέση που υπάρχει με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να καταλήξουμε σε ένα, ε, σε ένα φιλόδοξο κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών. Αυτός ο κατάλογος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ε, αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη τους καταλόγους αυτούς για την αναπτυξιακή πολιτική επίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει στη δημιουργία διαφανών ε, επιγραμμικών ε, μητρών ε, για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν στις χώρες αυτές και μας δυσχεραίνουν την αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλελεύθερη. Η Μάιτε Παγάσα Ορτοντού Ερουίθ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κάθε φορά βελτιώνεστε. Ε, Στη μέρα της ψηφοφορίας θα είστε τέλειος στην προφορά του ονόματός μου. Τα μαθαίνω, μαθαίνω. Μέχρι το τέλος της εντολής μας θα το έχω μάθει, ναι. Λοιπόν, οι συνάδελφοι προλαλήσαντες είπαν πράγματα που με κάλυψαν και εγώ τα ίδια κάπου θα έλεγα. Έχουμε μάθει πάρα πολλά αυτούς τους μήνες και ακόμα και αν τελειώνει η εντολή μας, η δουλειά δεν τελειώνει. Εκρεμούν ακόμα πολλά και στους συντονιστές γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Τι θα μας πούν οι πολιτικές ομάδες έτσι ώστε να δοθεί κάποια συνέχεια. Μόνιμη όμως συνέχεια να δίνεται. Γιατί τώρα που ζητήσαμε όλα αυτά, που μάθαμε όλα αυτά, δεν μπορούμε να την πετάξουμε όλη αυτή την εμπειρία. Κάτι πρέπει να γίνει. Ε, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και η Γραμματεία και το Προεδρείο και οι συγητές. Εξαιρετική σύντομα να πω μερικά πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να τερματιστεί η φορολογική αμνηστία, γιατί αυτό βοηθάει τα κράτη-μέλη να ε, κάνουν κακές πολιτικές. Δεν έχουμε κυρώσεις, κατάφορη απουσία κυρώσεων ε, παντού στα κράτη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λίστες ε, αλλά και κυρώσεις τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και επίσης μη συνεργαζόμενα κράτη, τις λεγόμενες δικαιοδοσίες που είναι πρόθυμες για συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε την εφαρμογή, ούτε τα ποιοτικά στοιχεία ε, των ε, οδηγιών για την καταπολέμηση του ξεκλήματος. Άρα πρόκειται για επένδυση εδώ. που θα έχει επιπτώσεις. Φυσικά χρειάζεται αυτόματη ε, ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Αλλιώς δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τη φορολογική απάτη και το ξέπλυμα. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα σύστημα άριστα ε, καταρτισμένο και ε, διαρθρωμένο για το ξέπλυμα και οι δικές μας ασπίδες είναι διάτριτες. δεν το είπανε πολλοί. Εταιρείε όπως είναι ιδιωτικέ τράπεζες, δικηγόροι, διαχειριστές, χαρτοφυλακίων, ιδιώτες κτλ. οργιάζουν. Έχουμε και άλλη λίστα εμείς, λίστα εκείνων που αρνήθηκαν να έρθουν να συνεργαστούν. Και έχουμε και μια αδυναμία γιατί στην ΑΦΚΟ το Συμβούλιο έχει ε, επανειλημμένα ε, βάλει τρικλοποδιά στην Επιτροπή μας γιατί αλλιώς θα είχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες. Λοιπόν, τα θεσμικά όργανα, διάφοροι φορείς, θεσμοί, ιδιώτες θα πρέπει να αντιδράσουν. Έχουμε προβλήματα, ξέρουμε ποια είναι, δεν μπορούμε να τα ε, αποφεύγουμε ή να ε, τα παρακάμπτουμε γιατί γνωρίζουν και οι πολίτες ότι υπάρχουν παραθυράκια και τρύπες, όχι μόνο παραθυράκια, γιατί διέρευσαν αυτά τα πράγματα και μας άνοιξαν τα μάτια. Ε, θα πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών γιατί αλλιώς αυτό συνιστά δυναμία δικιά μας. γιατί το συμβόλαιο το δημοκρατικό που έχουμε με το λαό και τους πολίτες. Είναι καταπληκτικοί οι ε, συγητές, το είπαμε, πολύ ενδιαφέρουσες οι τροπολογίες και ελπίζω να βγει τελικά μια θαυμάσια έκθεση και πολύ καλές συστάσεις. Αλλά, αλλά για να τελειώσω θέλω να πω και το εξής. Δεν έχουμε αξιόπιστες στατιστικές για το μέγεθος της φόρο-αποφυγής και φόρο-διαφυγής και αυτό πόσο επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στοιχεία ε, που έχουμε ακούσει, ξέρω εγώ, γενικά και πάρα πολύ αόριστα, δεν είναι συγκεκριμένα. Ε, Επίσης κάτι άλλο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την ομοφωνία στο Συμβούλιο για να νομοθετήσουμε για φορολογικά θέματα. Υπάρχει αυτή η σύσταση της Επιτροπής μας και αν δεν γίνει αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσουμε την κατάσταση αυτή. Ωραία τα λόγια, αλλά θα πρέπει να μεταφραστούν και σε πολιτικές και σε έργα αποτελεσματικά. Άρα, ένα νέο κέντρο συντονισμού και συνεννόηση της φορολογικής πολιτικής μπορεί να είναι ένα καλό βήμα προόδου. Δεν έχουμε καλές πληροφορίες, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ε, φορολογικές και για να αποθαρρύνουμε τη φοροδιαφυγή ε, θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Αυτό είναι ένα καλό αντικίνητρο για να μην φόρο αποφεύγει ή φόρο διαφεύγει με εταιρεία που θέλει να πάρει έργα. Επίσης έχουμε και τα πορίσματα της Επιτροπής Τάξε 1 ε, για ένα οργανισμό, ένα σημείο που θα γίνονται καταγγελίες. Η δουλειά δεν τελειώνει εδώ, μπορεί να τελειώνει δικιά μας. Ευχαριστώ ε, συνάδελφε Μάιτε. Και τώρα Γκουε. Ο Φάμπιο Μάζει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω και πάλι τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, ε, τους εισηγητές, συντονιστές, γραμματεία, και τους συνεργάτες των πολιτικών ομάδων για την ευχάριστη συνεργασία. Ακόμα και αν δεν συμφωνούσαμε πάντα πολιτικά, είχαμε πάρα πολύ καλή προσωπική σχέση με πολλούς συναδέλφους και λυπάμαι λίγο που φεύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν μπήκα στο Κοινοβούλιο είχαμε τα σκάνδαλα LuxLeaks, λίγο αργότερα τα έγγραφα του Παναμά και τώρα βάζω δημόσια ένα στοίχημα πριν φύγετε εσείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν ολοκληρωθεί η θητεία, θα αποκαλυφθούν και άλλα leaks και άλλες διαρροές θα έχουμε ε, για θέματα φορολογικά. Και αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε όλοι μαζί στην πλάση και θα σας κεράσω τηγανιτές πατάτες, όλη την Επιτροπή. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να βελτιώσουμε με την έκθεσή μας τι προτάσεις, να βελτιωθεί η νομοθεσία εκεί που δεν είναι επαρκή. Άρα, θεωρώ ότι έχει σημασία και θα φροντίσω και στη γερμανική βολή, στην Bundestag, να ελέγχουμε την κυβέρνηση και να τα εφαρμόζει όλα αυτά μια κυβέρνηση ε, του ΕΛΚ των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων και θα σας ενημερώνω κιόλας. Γιατί η δική μου πολιτική ομάδα έχει σημασία αποφασιστική στην οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος, να μην ε, ε, υπολοιπόμεθα τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ε, τριμερή διάλογο, δηλαδή να κλείσουν τα παραθυράκια για τους διευθυντές, για τα καταπιστεύματα, για τους πραγματικούς δικαιούχους και όλα αυτά τα δικήματα και να έχουμε και κυρώσεις. Εάν τράπεζες, δικηγόροι, λοιποί μεσάζοντες, ε, βοηθούν ε, την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και τη διευκολύνουν. Παράδειγμα, είχαμε μια ε, εκτίμηση της Μπάφιν στη Γερμανία που το μελέτησε αυτό και καταλήγει ότι παρά τα έγγραφα του Παναμά δεν είχαμε συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας. Δηλαδή όλα αυτά έχουν γίνει νόμιμα. Ε, άρα τα πρόστιμα και οι κυρώσεις ήταν πάρα πολύ χαλαρά στο παρελθόν και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η ομάδα ε, για τον κώδικα δεντολογίας αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Νίντερ Μάγια. Ξέρουμε ότι ακόμα και οι διπλωμάτες αναφέρουν στα πρωτόκολλα τους ότι δεν λειτουργεί καλά αυτή η ομάδα. Και χαίρομαι, αν υπάρχει εδώ πραγματική συνένεση, ε, να μην ξαναπέσουμε πίσω από τη θέση της τάξη 1 και να τα λέμε με το όνομά τους έχω την αίσθηση και το λέω με ε, συγκρατημένη ε, αισιοδοξία ότι θέλατε στη συνεδρίαση των σκιωδών το να χαλαρώσετε λίγο τα του κώδικα δεοντολογίας. Ε, η πολιτική μου ομάδα δεν το θεωρεί σωστό αυτό και θα γελιοποιηθούμε. Ακόμα και οι ίδιοι διπλωμάτες λένε ότι δεν πάει καλά αυτό. Φανταστείτε πόσο κακό θα ήταν να το αποδυναμώσουμε. Τα κριτήρια του μηδενικού φόρου για τις μαύρες λίστες. Αυτό το κριτήριο λέει δεν αρκεί για να εγγραφείς στον κατάλογο. Μα εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω στον κόσμο γιατί δεν θεωρείσαι φορολογικός παράδεισος όταν έχεις 0% συντελεστή εταιρικού φόρου. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Επίσης, το Accountancy Europe, που είναι ο Πανευρωπαϊκός Σύλλογος Ορκωτών Λογιστών και Οικονομικών Ελεγκτών, έχει κάνει τρομερό λόμπι ε, και έχει επικρίνει και τους σοσιαλιστές και τη δική μου πολιτική ομάδα και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα, τους πατήσαμε τον κάλο και ε, εμείς έχουμε αναθέσει και μια ε, μελέτη από τον Ρίτσαρτ Μέρφυ που ήταν ο ίδιος ορκωτός λογιστής και είπαμε ότι θα πρέπει να διαχωριστεί η παροχή συμβουλών ε, από την ε, ε, δικηγορική συνδρομή και τη βοήθεια για φορο απαλλαγή. Και μιλήσαμε για ευρωπαϊκή άδεια που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι λογιστές. Και θα ήταν κρίμα να περάσουν στην έκθεση οι τροπολογίε και επιθυμίες για αλλαγέ ε, αυτή τη οργάνωση που είναι λόμπι. Λοιπόν, ζήσαμε όλα αυτά τα σκάνδαλα και αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιωθούν οι αρμοδιότητε και εξουσίε του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν έχει να κάνει με κομματική τοποθέτηση που ανήκει ο καθένα, έχει να κάνει με το κύρο και τη φήμη του Κοινοβουλίου ω θεσμό. Άρα ε, πρέπει να έχουμε μια μόνιμη φορολογική ε, Επιτροπή. Γιατί σας έβαλα στοίχημα προηγουμένως, θα ακολουθήσουν και άλλα leaks. Να το ζητήσουμε και να έχουμε ένα ειδικό δικαίωμα κλήτευση των μαρτύρων να έρχονται εδώ να καταθέτουν και αυτοί που δεν συνεργάστηκαν, εδώ η Κατερπίλα και λοιπά, Μόνσακ Φονσέκα, ακούστηκαν τα ονόματα, να βρεθεί μια σαφής απάντηση γιατί αλλιώς πραγματικά και ε, αν δεν έχει συνέχεια αυτή η άρνηση για προθυμία συνεργασία και αν δεν έχει και κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τα άλλα, εύχομαι στην Επιτροπή μας ε, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και θα τα παρακολουθώ από τη Γερμανία αυτά με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, Φάμπιο Ντιμάζη. Σύντομα, δύο παρατηρήσεις για δύο θέματα. Για το μηδενικό φορολογικό συντελεστή, σύμφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι επίμαχο το θέμα, διότι ιδιαίτερα 35 συνολικά κράτη Ε, έχουν, υπάρχουν 35 μέρη που και στα, και στα κράτη-μέλη ε, με μεταβατικές διατάξεις, με προσωρινές διατάξεις όπως είναι η Μαδέρα και τέτοια ε, που έχουν μηδενικό φορολογικό συνδεδιστήριο που είναι φορολόγητα. Εγώ θα, θα ζητήσω να αλλάξει ακριβώς γι' αυτό. Γιατί εδώ ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιόνκερ είπε ότι κατά την άποψή του στην Ευρώπη δεν έχουμε φορολογικούς παραδείσους αν τηρούν όλοι ε, ε, τις νομοθεσίες. Αυτά δεν ε, ισχύουν, ε, δεν παληθεύονται από τα όσα μάθαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Είμαι όλοι σκοτκάτω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους και εισηγητές στις ευχαριστίες τους προς τους βασικούς εισηγητές Πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι απλώς τυπικότητα εδώ όπως συνήθως, το εννοούμε. Τεράστια δουλειά και επίσης ευχαριστίες προς τους συνεργάτες και τη γραμματεία. Διότι πραγματικά ε, φαινόταν ε, αδύνατο να τηρήσουμε την προθεσμία και συγχαρητήρια που τα καταφέραμε. Νομίζω η ποιότητα της δουλειάς αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι έχουμε τόσο σαφείς συστάσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε ευρία πλειοψηφία υπέρ Τη έκθεση ή δυνατόν απόλυτη στήριξη, διότι αυτό που θέλουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν ε, ε, παραμείνει σκανδαλισμένοι από την απουσία απάντηση ε, στα σκάνδαλα φοροδιαφυγής και πάτη που διαρκώ γνωρίζουμε. Πρέπει να δείξουμε λοιπόν ότι στο Κοινοβούλιο είμαστε ενωμένοι και αποκρινόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ότι είναι καλή συνεργασία με την Επιτροπή και ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι στο επίπεδο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο υποτίθεται ότι εκπροσωπείται στου ίδιου πολίτε που εκπροσωπούμε και εμεί, όμω ε, είμαστε θύματα αυτού του παιχνιδιού που παίζεται διαρκώ των παιχνιδιών ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Και αυτό δυσκολεύει την δυνατότητά μα να κάνουμε δημοσίω έρευνε. Πρέπει λοιπόν ε, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα, εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο για να αναλάβει δράση. Πρέπει να είμαστε επιτέλου αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Επίση, είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία και οι συστάσει μα να είναι σαφεί, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν επιτυχώ. Είναι δική μα ευθύνη να εκφράσουμε λοιπόν συστάσει με απόλυτη σαφήνεια και αν το κάνουμε αυτό μπορεί να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα πολιτικά θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε τη δημοκρατία να πιέζεται στον κόσμο μα. Και οι πολίτες διαρκώς ε, αμφισβητούν τους πολιτικούς και την πολιτική. Μπορούμε λοιπόν τώρα να δείξουμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και μπορούμε να βελτιώσουμε τις δουλειές τους τις ε, ζωές τους. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία βέβαια δεν συμφωνήσαμε απολύτω και ήθελα να τονίσω και την σκοπιά των πρασίνων. Πρώτα απ' όλα τα ευρήματα της έκθεσης ε, καθιστούν σαφές ότι όταν υπάρχει παραβίαση της οδηγίας για την, κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ε, βάσει των όσων έχουν αποφασίσει τα πολιτικά θεσμικά όργανα θέλουμε να είναι σαφές ότι αποφαινόμαστε για την μη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή και την ελληπή της υλοποίηση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη κάποιοι κανόνε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο που βρίσκονται σε διαπραγματεύση. Επίση για την αρχή του κατονομάζει και πονιδίζει. Εδώ ω Βρετανοί πολίτε πιστεύω για τι επικρίσει κατά τι αρχέ αυτέ. Ε, πολύ καλά γνωρίζω τους φορολογικούς παραδείσους ε, στην ε, χώρα μας και ξέρω ότι πολλές εταιρείες ε, που ε, είχαν ε, εμφανιστεί στα σκάνδαλα του Panama Papers, είχαν καταγραφεί στις Βρετανικές Παρθένους νήσους, Παρθένους νήσους και βάσει της Βρετανικής νομοθεσίας. Τα δικά μας λοιπόν, ε, οι δικές μας περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, μπορεί να είναι κέντρα φοροδιαφυγής. Είμαι απογοητευμένη λοιπόν με τις πρακτικές της ίδια μου τις χώρες, αλλά δεν πρέπει να διστάζουμε να κατονομάσουμε τι χώρε, ε, όσο κοντά μα κι αν είναι, που έχουν ε, εφαρμόσει αυτέ τι πρακτικέ. Βλέπουμε τώρα ποιε χώρε ήταν βασικοί παράγοντε ώστε να δώσουν τη δυνατότητα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Πρέπει να δούμε ότι υπήρξαν και οι ενδιάμεσοι που ήταν ο συνθετικό κρίκο όλο αυτό το μηχανισμό του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Μια έκθεση που ξεκίνησε ε, φέτο, την αρχή τη χρονιά, έδειξε τον σημαντικό ρόλο των ε, ε, ενδιαμέσων δικηγόρων ή τραπεζών που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στι περιπτώσει ε, φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Πολλέ φορέ βοήθησαν, ήταν υπεύθυνοι για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο. Λόγω λοιπόν αυτού του συσχετισμού, ξέρουμε ότι οι παραγόντε αυτοί εθελοτυφλούσαν στι πρακτικέ φοροδιαφυγή ή μπορεί να έχουν επιτρέψει σε πλουτοκράτε που ξεπερνούν τα εθνικά όρια να μην πληρώνουν καθόλου φόρο, όπως θεωρούν αυτοί ότι είναι σωστό. Ε, Είδαμε τα πρόσφατα ε, περιστατικά της Σλοβενίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και άλλα σκάνδαλα θα ανακύψουν. Γι' αυτό η θεσμική μας απόκριση πρέπει να είναι κατάπαυστη. Πρέπει να συνεχίσουμε να διερευνούμε τα θέματα αυτά. Είναι σημαντικές οι συστάσεις μας, διότι αν δεν βεβαιωθούμε ότι υπάρχει εξακολούθηση και προσοχή στο πώς υλοποιούνται, δεν έχει νόημα. Χρειάζεται λοιπόν και μια αυτή η τροπολογία που να βεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να οργανώσει μια μόνιμη εξεταστική επιτροπή για τα θέματα αυτά Κάτι που ούτω ή άλλω αποτελεί σύστημα νομιμοποιημένο στι ΗΠΑ μέσα τη γερουσία. Πρέπει λοιπόν τα σκάνδαλα ξεπλήματο βρώμικου χρήματο ε, να βασίζονται στην διερεύνηση εγγράφων, τα οποία να έχουμε δικαίωμα να ζητούμε με κάποια ε, κλήτευση ή με ε, ένταλμα. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η φορολογική πολιτική διερευνά τα φορολογικά σκάνδαλα για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη. Και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι συστάσει μα που σαφώ έχουν διατυπωθεί υλοποιούνται κιόλα. Ευχαριστώ πολύ, Μόλι. Ο Ντέιβιτ Κόμπορν, ε, τελευταίος εκπρόσωπος πολιτικής ομάδας και μετά ο Τόμα Μάν. Uh, danke, Herr President. Um, ε, two reports that this committee οι δύο εκθέσεις που θα εγκρίνει η Επιτροπή μας, όπως και οι τροπολογίες, δείχνουν ότι ε, ακόμη είμαστε εργοστάσιο παραγωγής ε, νομοθεσίας, ότι έχουμε λίγο σεβασμό για τον ιδιωτικό βίο, λίγη κατανόηση της επιχείρησης, των επιχειρήσεων και του εμπορίου, όπως επίσης και του πλούτου που δημιουργούν οι ιδιώτες και οι εταιρείες. Ε, αυτό κυρίες και κύριοι θα είναι επιβλαβές ε, και για, την, ε, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και για την απασχόληση γιατί θα σκοτώσετε τις επιχειρήσεις, θα τις στραγγαλίσετε, όπως επίσης και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομική ανάπτυξη που ήδη βλέπουμε σήμερα. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλο ιστορικό ε, καταστροφή των επιχειρήσεων λόγω των ε, ρυθμίσεων που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Γι' αυτό ε, οι Βρετανοί αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. η Μεγάλη Βρετανία Γερμανία και το ε, City ε, δυστυχώς ε, κρατούνται δέσμοι ε, με, λόγω των ε, ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο σκοτώνει ε, τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες, κάτι το οποίο νομίζω είναι ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τέρας το οποίο καταπίνει όλο και περισσότερο χρήμα για να πληρώνει όλο και περισσότερους γραφειοκράτες. Και αν δει ε, αν κανείς καταστρέψει όλους τους τρόπους μείωσης των ε, φόρων, τότε γιατί να δίνουμε τα <laughs> χρήματα ε, σε κυβερνήσεις που τα ξοδεύουν σε διάφορα γελία πειράματα στις περιφέρειες Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παραδειγμα και να, καλέ, να ακολουθήσουν κι άλλοι στην εγκατάλειψη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως η Καταλωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ε, αθέμητο, τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό. Συγγνώμη. Και εκεί είναι πρωταθλητή η Μεγάλη Βρετανία δυστυχώ. Όχι μόνο ε, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατία. Ε, εντάξει, είναι ανθρώπινη αδυναμία αυτό και ιδιότητα να μην θέλει κάποιο να πληρώνει φόρου, γιατί το πιο ευαίσθητο μέρο του σώματο ακόμα παραμένει το πορτοφόλι. Είναι ανθρώπινο δικαιώμα να διατηρείς τα λεφτά σου. Να πρέπει να, να επιβραβεύεται ο, η σκληρή δουλειά και όχι η γραφειοκρατία που πνίγει τον κόσμο. Και αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Μεγάλη Βρετανία θα δώσει παράδειγμα στον κόσμο οικονομικής αποτελεσματικότητας και πώς πρέπει να γίνεται αυτό είναι δικαίωμα του κάθε πολίτου τα λεφτά που βγάζει με τον υδρότα του να μπορεί να τα κρατάει. Έχει δουλέψει σκληρά και όχι να τα δίνει σε μερικούς γραφειοκράτες που απλώς του ρουφούν το αίμα. Καλά, θα δούμε πώς θα πάει το Brexit. Ε, Επόμενοι ε, λοιποί ομιλητέ, ο Τόμας Μαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλες οι τοποθετήσεις ε, που ακούσαμε μέχρι τώρα ε, ε, έπονταν από κάποια νοσταλγία εκτός από την τελευταία ε, που ήταν γεμάτη κλισέ. Να δώσουμε ένα φυλάδιο στον συνάδελφο να το εξηγούμε τι είναι η κοινωνική οικονομία τη αγορά. Κοιτάξτε, εμεί είμαστε εξεταστική επιτροπή και όχι ειδική έκτακτη επιτροπή. Καλό είναι αυτό. Έχουμε πολλέ αρμοδιότητες και συμφωνώ και με την ιδέα του Φάμπιου. Τον ευχαριστώ για όλη αυτή τη συνεργασία αυτά τα χρόνια. Δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά από την αρχή ε, είχαμε πολύ ποιοτική σχέση και συνεργασία. Καλό είναι λοιπόν να πούμε ε, να έχουμε ένα δικαίωμα κλήτευσης μαρτύρων ή να φροντίσουμε να υπάρχει μια μόνιμη φορολογική επιτροπή γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ε, σοβαρό γιατί διακυβεύεται η αξιοπιστία μας. Πώς θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα δύσκολα και τα κακό σκήμενα. Με λόγια, όχι, με έργα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και ελπίζω και οι συμβιβασμοί να πάνε προς την κατεύθυνση αυτή και να ζητούν κυρώσεις για εκείνους που δεν ε, ε, ήρθαν. Σωστά είπε Λόγκεν ότι έχουμε διαφορές. Από τη μια έχουμε αυτή τη δημιουργική φορολογική αντιμετώπιση ε, που όπως είπε και ο εισηγητής αυτό είναι νόμιμο αλλά όχι ωραίο ε, και το άλλο είναι παράνομη φόρο αποφυγή. Αυτό το κάναμε τώρα. Ε, περιμένω τα αποτελέσματα των συμβιβασμών. Για μένα θα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε ο Ιούνκερ να υπογραμμιστεί όταν μίλησε για την κατάσταση στην Ένωση. Δηλαδή ότι υπάρχει ε, ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μα ακριβώς τα φορολογικά θέματα διαπιστώνουμε ότι παραμένει στην ομοφωνία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να περάσει στην ειδική πλειοψηφία. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε φορολογικές οάσεις και φορολογικούς παραδείσους στα κράτη-μέλη. Και ένα σημαντικό για μένα επίσης και η ψηφιοποίηση. Υπάρχουν ψηφιακές έδρες, εικονικές, που αιωρούνται κάπου στην ατμόσφαιρα. Δεν έχουν έδρα σε συγκεκριμένη χώρα, επικράτεια. Δίκαιο. Και αυτές οι εταιρείε ταχυδρομικές σειρίδες που υπάρχουν παντού έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μια ιδέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια ιδέα που εμείς την απορρίψαμε, τη σπάσαμε, την κόψαμε, να υπάρχει αυτομική εταιρεία προσωπική να μπορεί να ιδρύει κάποιος, να καταθέτει ένα ευρώ, αλλά χωρίς να έχει έδρα πουθενά. Δεν γίνεται αυτό. Και όταν έρθουν οι επόμενες περιπτώσεις και σκάσουν τα επόμενα σκάνδαλα, δεν θα πρέπει να λέμε τη δουλειά κάνουν οι δημοσιογράφοι και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να κάνουμε. Ε, με ε, καλό πνεύμα επικοδομητικό, με συνεργασία, με νομικά επιχειρήματα που να ευσταθούν και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί αυτή η δουλειά και για τους πολίτες να στεφτεί με επιτυχία η εντολή αυτή που μας έδωσε το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας Μαν. Τελευταίος Άλλους τρεις έχω δηλαδή, αλλά και οι τρεις είναι απόντες. Επόμενος, ο συνάδελφος Χάουρεγγι. Παρακαλώ, Ραμόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω και με τους δύο εισηγητές, το Γέπε και το Πέτερ, αλλά και το Προεδρείο. Κύριε Λάγκεν, πραγματικά το Προεδρείο έτσι με κάποια γερμανική τάξη καμιά φορά διεύθυνε τις συνεδριάσεις αλλά και με ανοιχτό πνεύμα ε, και ε, για να μπορέσουμε να φέρουμε εδώ όλους όσοι έπρεπε να έρθουν να καταθέσουν. Ε, Κοίταξτε, είναι σημαντικό το έγγραφο και θα ήθελα να τονίσω το εξή στους συναδέλφους. Δεν υπάρχει πουθενά κοινοβούλιο στον κόσμο. Καλά, το Βελγικό Κοινοβούλιο έχει κάνει κάποια δουλειά, αλλά τόσο εξαντλητική για το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο, σαν αυτό που έκαναμε εμείς. Και πραγματικά η δουλειά μας θα επιτρέψει, πιστεύω, ε, σε όλη αυτή την υπόθεση για φορολογική δικαιοσύνη να έχει ένα δικό χάρτη, ένα δρόμο, ένα φύλλο πορείας για να προχωρήσει. Εύκολο δεν θα είναι καθόλου να εφαρμοστούν τα διάφορα μέτρα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι χτίσαμε και φτιάξαμε αυτό που έλεγα ε, το οδόστρωμα. Δηλαδή έχουμε στρώσει αυτό το δρόμο τώρα και όπως είπε και ο Φάμπιο θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, δεν τελειώνει εδώ. Αλλά για την υπόθεση της φορολογικής δικαιοσύνης έχουμε ανοίξει ένα δρόμο. Και συμφωνώ και με τη Μόλη και με τον Φάμπιο κάτι πρέπει να υπάρξει ως συνέχεια. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο ποιος ε, θα είναι αυτό το σύστημα. Αλλά θα ήταν ωραίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα περισκόπιο έτσι βγαλμένο, ένα παρατηρητήριο και να επιθεωρεί και να συνεχίζει να παρατηρεί τα όσα συμβαίνουν. Έχω κάνει πολλές τροπολογίες και εγώ και η ομάδα μου προφανώς και αισθάνομαι ικανοποιημένος για όλα αυτά τα επιτεύγματα. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σας περι περιγραψω τρει τέσσερι ιδέες που πιστεύω ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί ε, αρκετά και το είπαν και κάποιοι άλλοι. Πρώτον, στην οδηγία της συνεργασίας που ισχύει τώρα θα πρέπει ε, να επεκτείνουμε τον κατάλογο εκείνων που υποχρεούνται να δίνουν πληροφορίες. Ε, στην οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος υπάρχει ένας κατάλογος διαφόρων φορέων που είναι σε αυτό το κύκλωμα το χρηματοπιστωτικό, αλλά στην οδηγία για τη συνεργασία όχι. Και είναι σημαντικό στη φορολογική συνεργασία να συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί οι παράγοντες, ε, συμβολεογράφοι, διάφορα γραφεία, πράκτορες, ε, διαχειριστές χαρτοφυλακίου, άλλες εταιρείες. Αυτά δεν τα λέει επαρκώς πιστεύω η έκθεση. Δεύτερο, ε, τα κράτη έχει σημασία να ε, θωρακιστούν κάπως ή να θωρακίσουν τις προσφορές που κάνουν ορισμένοι επιθετικές φορολογικές, γιατί πολλές χώρες κάνουν προπαγάνδα, όχι διαφήμιση, σε οικονομικούς χώρους και προσφέρουν ε, τους φορολογικούς ε, χώρους τους που είναι αρκετά αδιαφανείς και θολοί. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές διάδοσης, διαφήμισης ε, της φορολογικής θολούρας για να προσελκύσουν τα κεφάλαια είναι απαράδεκτες και θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Τρίτον, θα πρέπει να είμαστε πιο κατηγορηματικοί με τις εσωτερικές απαγορεύσεις στα ίδια μας τα κράτη-μέλη διαφόρων πρακτικών που ευνοούν τη φοροαποφυγή. Παράδειγμα, να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας των τραπεζών που βοηθούν. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η κύρωση να απαγορεύεται η συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείε που έχουν δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους, να αποκλείονται από τους διαγωνισμούς και σε φυσικά και οι νομικά πρόσωπα να μην επιτρέπεται να ανοίγουν ε, τραπεζικούς λογαριασμούς ή εταιρείε στις χώρες της μαύρης λίστας. Αυτό δεν εκφράζεται παρκώς κατά την άποψή μου. Ακόμα κι αν όλα αυτά είναι στόχοι που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν και να υιοθετήσουν, ε, είναι σημαντικό να μην χάσει η έκθεσή μας το χαρακτήρα της του ε, καθολικού οδικού χάρτη για να έρθουν τα κράτη να τα εφαρμόσουν. Και ένα ίσονος ίσως σημασίας μέτρο, αλλά για μένα είναι σημαντικό η Ευρώπη να εναρμονίσει την Ε, μάλλον το ποσό που μπορεί κανείς να χειρίζεται σε μετρητά. Δηλαδή, στη Γαλλία απαγορεύεται να πληρώνεις ένα ποσό άνω των χιλίων ευρώ με μετρητά. Αυτό είναι καλό μέτρο που ε, βοηθάει και την καταπολέμηση της φοροδιαφύγης και δεν το γράφει η έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσει την ευκαιρία να πω τις ιδέες μου αυτές που θα τις διατηρήσουμε σε κάποιες τροπολογίες και θα τις ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Καλώς. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και έχουμε διάφορες προτάσεις για τη χρήση μετρητών. Υπάρχουν και διαφορετικές παραδόσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει να το δούμε στην κανονική νομοθετική διαδικασία ξεχωριστά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικό στο να περιορίσει γενικά τα μετρητά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπει στη παρούσα έκθεση. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Τώρα, η Άννα Γκόμες, η οποία εδώ ήταν, αλλά πήγε να ψηφίσει που ψηφίζουν στην Επιτροπή Λίμπε, αν δεν απατώμε. Έχω το συνάδελφο Φαντεκέντελαρ που είναι σε άλλη επιτροπή και ψηφίζει. Αυτά είναι όταν συνεδριάζουν ταυτόχρονα οι επιτροπές. Οπότε θα δώσω το λόγο. δεν θέλει κανένα άλλο. Δεν θυμάμαι, σήκωσε κανένα κανένα χέρι. Α, κύριε Κόμπορν. Μην κάνετε τώρα δήλωση από τι αρχέ. Κύριε Πρόεδρε, απλώς αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο κύριος, ε, για την περιορισμό των, ε, της χρήσης των ρευστών. Κοίταξε, αυτό είναι τεράστια παρεξήγηση και δεν υπάρχει κατανόηση καμίας μορφής επιχείρηση Πώς μπορεί να λέει κάτι τέτοιο. Προφανώ δεν έχετε καμία ιδέα περί τίνο πρόκειται, τι είναι η επιχείρηση. Αυτή η πρόταση είναι γελία πραγματικά. ja, das gibt's auch. Καλά. Αυτό υπάρχει και σε χώρες και επικράτειες που είναι υπό τη Βρετανική επιρροή. Στην Τουρκία, α πούμε, αν πάτε και πείτε τέτοιο πράγμα, θα σα κοιτάνε με γουρνωμένα τα μάτια. Ε, σε άλλε χώρες που είναι πιο κεντρικά δικούμενες ε, αυτό μπορεί να ισχύει. Θα δώσω το λόγο ξανά στον κύριο Χάουρεγγι. Κοιτάξτε, ήθελα να πω στον συνάδελφο μόνο ότι αν έβλεπε ένα χάρτη της Ευρώπης και κοίταζε και εξέταζε τι απαγορεύσει εχουν έχουν επιβάλει κάποια κράτη-μέλη ήδη στην κυκλοφορία των μετρητών. Για τα ποσά δηλαδή που συζητάμε θα ανακάλυπτω ότι αυτό που λέω δεν είναι καμιά ανοησία. Περίπου 12 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη περιορίσει το ποσό. Μεταξύ αυτών και η Γαλλία. Και στην αγορά ε, ε, λειτουργούν οι γαλλικές εταιρείες, δεν είναι και τίποτα ηλίθιοι. Άρα, στη γραμμή αυτής τη έκθεση θα έλεγα, που εξετάζει δρόμους για να προχωρήσουμε, θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίσει το ποσό που επιτρέπεται να διαχειρίζεσαι σε μετρητά. Ισχύει όμως ήδη σε πάνω από 12 ευρωπαϊκές χώρες, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος αλλά μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Οι εγκληματίες δεν χρειάζονται μετρητά πια, ε, ιδρύουν εταιρεία ή ακόμα και τράπεζα για να οργανωθούν έτσι, δεν χρειάζεται να κυκλοφορούν τα μετρητά. Οπότε και η κατάργηση του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί σταμάτησε να τα τυπώνει μπορεί να είναι σκόπιμο και λογικό αλλά δεν υπάρχει ε, νομίζω πλειοψηφία στην Ευρώπη για τον περιορισμό των μετρητών. Αν δεν θέλει κανένα άλλο λόγο, ε, ε, ε το λόγο, συγγνώμη, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Thank you so much, uh, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις πολύτιμες συνεισφορές τους ο Λίντερ Μίντερμα δεν είναι τώρα εδώ, αλλά είπε στην αρχή της παρέμβασής του ότι είναι σημαντικό η έκθεσή μας να είναι πλήρης και μια καλή ε, συμβαστική λύση. Έμπνευση ε, για, πηγή για περαιτέρω δουλειά. Και το λέω από την αρχή γιατί σε κάθε περίπτωση και από αυτή την πλευρά ακούστηκε ότι γενικώς Κάποια πράγματα καλά είναι στην έκδοση, αλλά πρέπει να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Είναι πολλές οι αυτές οι πτυχές. Σίγουρα είναι μια νέα δομή αυτή που έχουμε δημιουργήσει εδώ, αλλά και σε άλλες επιτροπές και δουλειές του Κοινοβουλίου θα πρέπει όλες αυτές οι συστάσεις να λαμβάνουν υπόψη και να ε, εφαρμόζονται. Επίσης, για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη, τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικέ στρατηγικέ κατά των δύο φαινομένων. Αν πάρουμε την φόρο αποφυγή, τη φόρο μάλλον, χρειάζεται περισσότερη επιβολή του νόμου, χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν αυτός, ό,τι αφορά την αποφυγη πρέπει να αντιδράσουμε και εδώ κάπως, ότι οι φόροι πληρώνονται και ότι υπάρχει κέρδος και κερδοφορία. Ότι με όλη αυτή τη λιτότητα που επικρατεί δεν υπάρχει άδικο φορολογικό ανταγωνισμό και ότι ζημιώνονται οι κοινωνίε μα. Πρέπει και τα δύο λοιπόν να πηγαίνουν παράλληλα. Πρέπει ε, μέσα από τη συζήτησή μα να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ στρατηγικέ κατά των δύο φαινομένων που μπορούν να εφαρμοστούν. Ε, ακούστηκε και το είπα και στην συνάδελφο από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, ε, τι θα γίνει με κάποιε εταιρείε, ε, τι εικονικέ εταιρείε που είναι απλώ δομέ ε, είναι οντότητες απλώς, νομικές, νομικά πρόσωπα ή κενές ε, περιεχομένου. Εάν κάποιος όμιλος ή κάποια εταιρεία ε, έχει αρκετά χρήματα, μπορεί να, αγοράσει, να εξαγοράσει την ανωνυμία και να χρησιμοποιήσει αυτή τη δομή για παράνομους σκοπούς. Αυτό είναι κάτι που το διαπιστώσαμε πέρα αμφιβολίας. Πρέπει να πω κάτι λοιπόν ανεξαρτήτω πολιτική ομάδα ότι όλοι ανέφεραν έναν κώδικα συμπεριφορά για την φορολόγηση των εταιριών και το μέρο του Συμβουλίου, το ρόλο του Συμβουλίου σε όλη αυτή την εξίσωση. Συμφωνώ. Υπάρχει ένα αγώνα που πρέπει να ε, ασκηθεί για την πίεση που θα, ε, θα ασκήσουμε προ το Συμβούλιο για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή ω πηγέ χρηματοδότηση μέχρι και τη τρομοκρατία. Κάτι πρέπει να γίνει. Ένα κώδικα λοιπόν ε, συμπεριφορά για την φορολόγηση των εταιριών, κάτι που εδώ και 19 χρόνια θα έπρεπε να έχει επιληθεί για να ε, αντιμετωπιστούν οι φορολογικές, οι φορολογικοί διακανονισμοί, οι διμερείς φορολογικοί διακανονισμοί μεταξύ κρατών δεν μπορεί να είναι κάτι που θα συνεχιστεί για πάντα. Υπάρχουν εταιρείε που λειτουργούν εκτό τη δημόσια σφαίρα ε, ΣΑΗ. Ε, εδώ και καιρό μάλλον. Και πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα μπορούσε αμέσω να περάσει σε μία πραγματική αξιολόγηση του ότι έχει γίνει τα τελευταία 19 χρόνια για τον κώδικα συμπεριφορά για την φορολόγηση των εταιριών. Κατά πόσον ε, οι επιζήμιες διακρατικές ε, φορολογικές αποφάσεις ε, έχουν πετύχει το στόχο τους ή όχι. Και το Συμβούλιο θα έπρεπε να αλλάξει τη στάση του. Ξέρω ότι οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν περισσότερη διαφάνεια όταν συζητάμε τέτοια ζητήματα. Και πρέπει να δούμε ποιε είναι οι χώρες, ποιε είναι οι κυβερνήσει που μπλοκάρουν αυτές τις αποφάσεις. Είναι λοιπόν σαφής η ανάγκη για μεταρρύθμιση. Έγιναν πολλά σχόλια, όπως είπα, Το θέμα των καταλόγων, ε, η συμμόρφωση, οι κυρώσεις, ε, ο μαύρος κατάλογος. Το σημαντικό δεν είναι στο τέλος να έχουμε απλώς ένα κατάλογο, αλλά να έχουμε και πραγματικές κυρώσεις για να πιέσουμε κάποιοι να αλλάξουν την ε, συμπεριφορά τους, τη διαγωγή τους. Να λαμβάνουν υπόψη τα πρότυπα και να τα εφαρμόζουν. Πρότυπα που είναι απαραίτητα για να καταπολεμηθούν φορολογικοί παράδειση λόγου χάρη. Συμφωνώ λοιπόν κατά πολύ με αυτό. Επίση υπόθηκε από αρκετού συναδέλφου, από την Άλντε λόγου χάρη, ότι εν τέλει πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μα. Την εμπιστοσύνη στο ε, στα θεσμικά όργανα και στο κοινωνικό συμβόλαιο, όπως ε, είπε κάποιος άλλος συνάδελφος. Ναι, Κάποιοι καταφέρνουν να πληρώνουν μηδέν φόρους σχεδόν. Ή όταν ε, πρόκειται για μεγάλε πολυεθνικέ, ε, τι μεγάλε τεχνολογικέ εταιρείε, πλέον σχεδόν 0% φόρο. Ενώ οι μικρομεσαίε έχουν φορολογικό βάρο πολύ μεγαλύτερο από ότι οι μεγάλε πολυεθνικέ. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Δεν είναι δίκαιη η οταν προκειται για μεγαλες πολυεθνικες τις μεγαλες τεχνολογικες εταιρειε πληρωνουν σχεδον 0 φορο ενω οι μικρομεσαίες εχουν φορολογικο βαρος πολυ μεγαλυτερο απο οτι οι μεγαλε πολυεθνικε δεν ειναι δικαιο αυτο δεν ειναι δικαιη η κοινωνια αυτη Και το βλέπει ο κόσμος. Το βλέπει ότι οι πλούσιοι, οι διασημότητες, οι αστέρες του ποδοσφαίρου και το καθεξή, ε, φοροδιαφεύγουν. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, εάν με επιτρέπετε, το όλο θέμα της εξακολούθησης, της συνέχεια που θα δοθεί, είναι καθοριστική σημασίας να καταλάβουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, η Φιλανδή συνάδελφος από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Η δουλειά αυτή μόλι ξεκίνησε. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε με την έγκριση αυτή τη έκθεση. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει κάποια συνέχεια στην προσοχή που θα δοθεί στο όλο θέμα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με όλου. Δεν είναι απλώ το θέμα να καλύψουμε με τις συμβαστικές της μέρημνας όλο σε μια έκθεση. Πρέπει η δουλειά μα να συνεχιστεί. Ω προ το κατονομάζει και πονηδίζεν. Ε, πρέπει να πω για μένα ως εισηγητή είναι σημαντικό στα ευρήματά μας, στη δουλειά μας, να παραμένουμε πολύ ακριβείς ε, για όσα είδαμε και διαπιστώσαμε. Δεν υπάρχει κατονομάζουν και πονηδίζουν, αλλά αναφέρεται το ποιες ακροάσεις είχαμε, με ποιους συνομιλήσαμε, ποιοι δεν ήρθαν, ε, κατονομάζονται ε, και πονιδίζονται εφόσον δεν ήρθαν ως εδώ αλλά προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς και ε, σαφείς γινόταν μέσα από τη δουλειά μα. Και βεβαίως εταιρείε, δικηγόροι, ενδιάμεση, όποιοι έχουν παίξει κάποιο ρόλο ε, σε όλη αυτή την υπόθεση και γιατί ε, έδειξαν ενδιασμό να συμμετάσχουν στη δουλειά μα. αυτοί ε, καλώ αναφέρονται. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου και ευχαριστώ πολύ και εσά, Πρόεδρε, για την υποστήριξή μα σε αυτή την τόσο σημαντική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ και τη Γραμματεία για την υποστήριξή του και το λέω αυτό όχι μόνο εκ μέρου των συνεισηγητών, των δύο συνεισηγητών, αλλά όλων των πολιτικών ομάδων που συμμετείχαν στη δουλειά μα. Νομίζω ότι δείξατε ε, ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, ακόμη και με κάποιο ε, περιορισμένο νομικό πλαίσιο και περιορισμένου πόρου. Κάτι καταφέραμε με την τόσο καλή δουλειά τη γραμματεία και την συμμετοχή του Πρόεδρου. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ τον, ε, τον εισηγητή. Ε, αναφερθήκατε σε όλα τα σημεία που σημειώθηκαν προηγουμένως και χαίρομαι και για τους συμβιβασμούς που θα κάνουν διάκριση των ε, παρανόμων και των ε, νομίμων ε, δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν, που μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι πάντα ωραίο αυτό που ακούσαμε, αλλά είναι νόμιμο. Το είπε και συνάδελφο Μόλι Σκοτ κάτω και το σημείο σε αυτά είναι παιχνιδάκι των εταιριών. Δεν ισχύει αυτό. Οι εταιρείε εκμεταλλεύονται αυτό που τους επιτρέπουν τα κράτη-μέλη ή άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που προσφέρουν ως κίνητρα για να προσελκύσουν επενδύσεις και εταιρείε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία. Όπως είπε η Εύελιν Ρέγνερ, αυτό είναι ο σωστός δρόμος και όχι να κατηγορούμε ε, τις εταιρείες και στην ακρόαση της BASF ακούσαμε και ήταν ο υψηλότερος ε, μάνατζερ παγκοσμίω για τα φορολογικά που ήρθε και είπε ότι κοίταξαν δείτε εμεί εκμεταλλευόμαστε και αξιοποιούμε αυτό που προσφέρεται και το οφείλουμε αυτό και στους μετόχους μας να το κάνουμε. Άρα η πολιτική φέρει τον πρώτο και κύριο ε, ρόλο και την πρώτη ευθύνη. Ε, εδώ Είχα ακόμα τον Τόμ Φαντεκέντελάρε στον κατάλογό μου που άκουσε εδώ το, το συμπέρασμα. Είχε κλείσει ο κατάλογο των ομιλητών. Ζήτησα συγγνώμη για την απουσία σου γιατί ψήφισε, όπω και η συνάδελφο Αναγκόμε, σε άλλη επιτροπή. Α, ήρθε και ο κύριο Ρωσάτη τώρα. Δεν ξέρω, έχετε σχόλια αφού ακούσατε τον εισηγητή. Λίγο χρόνο ακόμα έχουμε. Η Μόλι και μετά ο Ντάριο Ρωσάτη be uh, Ναι. Νόμιζα ότι θα υπάρξουν δύο γύρες στη συζήτηση. Αλλά απλώς να επιστήσω την προσοχή σε κάποιες από τις ε, βασικές τροπολογίες μας που δεν συμπεριλήφθησαν στις ε, συμβαστικές και είναι σημαντικές για μας ε, ως ομάδα. Είμαστε σε ένα ταξίδι εδώ, σε μια διαδρομή και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι διανύουμε ένα δρόμο και κάποια πράγματα μπορούμε να τα ξαναβρούμε μπροστά μας την πορεία αυτή. για για τις εταιρείες, ε, για τις εικονικές ε, ε, εταιρείες και για μια πρόταση που καλό θα ήταν να υπάρχει εδώ. Θα πρέπει οι εταιρείε να παρέχουν κάποιο οικονομικό αιτιολογικό, ε, αιτιολόγηση για την προλογική δικαιοδοσία στην οποία υπόκεινται. Ε, τροπολογία 65. Λέει ότι το βάρο τη απόδειξη το έχουν εταιρείε και να λένε ότι έχουν οικονομικού λόγου για να αλλάξουν ε, την ε, φορολογική του έδρα και όχι μόνο για σκοπού φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Έπειτα ένα-δυο ζητήματα που έχουν να κάνουν με του και τα ανέφερα και προηγουμένω. Και είναι σημαντικά ως προς τις αθέμετες φορολογικές πρακτικές. Έχουμε την αρμοδιότητα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Κοινοβούλιο να κάνουμε κάτι εδώ. Πιστεύουμε ότι οι δικαιούχοι των ε, οικονομικών ε, ενδιαμέσων που έχουν συμμετάσχει στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Μεγάλα ποσά τους έχουμε δώσει και θα πρέπει να απαιτούμε αυτοί που τα λαμβάνουν να είναι στα υψηλότερα επίπεδα, επίπεδα εντιμότητας. Ε, αυτό δεν υπάρχει τελικά στην έκθεση και θα θέλαμε να ενισχυθεί κάποια στιγμή. επίσης, Ω προ του ενδιαμέσου, πιστεύουμε ότι δεν μπορούν οι ίδιοι να αυτορυθμίζονται. Πρέπει να υπάρξουν υψηλότερα πρότυπα κώδικε συμπεριφορά για του δικηγόρου και του λογιστέ. Θα πρέπει η αυτορύθμιση να συνοδεύεται από την απαραίτητη επίβλεψη και την κρατική ε, νομοθεσία ε, ή από μια ανεξάρτητη αρχή που θα ρυθμίζει ή θα επιβλέπει. Επί, όχι πολλά ακόμη, δυο μόνο. Η τροπολογία μας 177 ζητά από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, να την οδηγία της περί ε, δημόσιων προμηθειών, ώστε εταιρείε που έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιε. Και οι φορολογικές συμφωνίες να μην επιτρέπουν το εμπόριο με χώρες που έχουν επιτρέψει του φορολογικούς παραδείσους ή έχουν μυστική νομοθεσία. Οι τροπολογίε μα αυτέ θεωρώ ότι είχαν κάποιο νόημα και θα φροντίσω να τη στείλω με mail στου υπόλοιπου συναδέλφου για να ξέρουν και τι περιλήψει συμβαστικέ. Θέλω να διαφωνήσω ρητά σε ένα σημείο. Το δικαίωμα στην αυτορύθμιση των διαφόρων ενδιαμέσων γενικά έχει αποδειχθεί καλό. Είναι τμήμα ε, τη επίσημη νομοθεσία σε πολλά κράτη-μέλη. Εκεί που συμφωνώ είναι να υπάρχει υποχρέωση ε, αναφοράς και έλεγχος από τους κρατικούς θεσμούς. Άρα αυτό που λένε γενικά οι πράσινοι, να καταργηθεί η αυτορύθμιση από παντού, ούτε ρεαλιστικό είναι, ούτε μπορώ να το υποστηρίξω. Ο Ντάριος Ρωσάτη για δύο λεπτά και πάλι. Yes, thank you, Chairman. Ε, I apologize. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ήμουν στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας. Έπρεπε να είμαι πρόεδρος σε μια άλλη συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Θα ήθελα όμως δύο σημεία να επισημάνω. Καταρχάς εμείς στο ΕΛΚ πάντοτε ενδιαφερόμασταν για μια ισχυρή έκθεση που θα αποστείλει ένα σαφές μήνυμα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται κάποια δράση για να μπορέσουμε να μειώσουμε το μέγεθος του φαινομένου της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και του ξεπλήματος ε, χρήματος και υποστηρίζοντας ε, την έκθεση και το σχέδιο συστάσεων, πρέπει να πω ότι εντυπωσιάζομαι από το πόσο πολύ συμφωνούμε. Είχαμε δύσκολες συζητήσεις. Είναι πραγματικά εκπληκτικό που καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Και παρά το γεγονός ότι παραμένουν εκκρεμή ζητήματα, τα οποία όμως κατά τη γνώμη μου είναι ίσομνος σημασίας, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα εξομαλύνουμε και να συμφωνήσουμε κατά τις ερχόμενες ημέρες. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους δύο εισηγητές ε, για τη δουλειά τους και για την ε, θέλησή τους να συνεργαστούν με όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεύτερον, ζητήματα διαφιλονικούμενα όπως το κατονομάζει και πονηδίζει ο μαύρος κατάλογος, η συνέχιση των εργασιών μας. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μας ε, πρότεινε καλό συμβιβασμό, μπορούμε να το συζητήσουμε στις πολιτικές μας ομάδες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη τους υπάρχοντες φορείς όπως ε, η ομάδα εργασίας για τους, ε, για τους φόρους εντός Επιτροπής ΕΚΟΝ ή τις επιτροπές Γιούρι, Λίμπε και Έκον να συνεχίσουν ε, την παρακολούθηση του θέματος. Πάντως η δουλειά μας δεν πρέπει να σταματήσει μετά την εκπόνηση της έκθεσης. Πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα γιατί όλο προκύπτουν νέες ε, υποθέσεις ε, που πρέπει να εξεταστούν. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εξακολουθήσει να επαγρυπνεί ε, για να εξακολουθήσει να πιέζει και τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ώστε να καλύψουμε τα κενά αυτά και να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε σοβαροί ως προς τους φόρους, γιατί είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από μας να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γέπε, ε, κόφωτ σύντομα για να κλείσεις. Προς την ίδια πηγαίνουν νομίζω όλα αυτά. Και μετά να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Ναι. Πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Καταρχή, κατα, καταρχήν καταφέραμε να, υπάρξουν, να υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και να καλύψουμε τα ζητήματα που ετέθησαν σήμερα ε, και στα δύο κείμενα. Ε, με τους πολιτικούς συμβιβασμούς είμαι ικανοποιημένο. Μπορεί πάντοτε κάποιος να πει ότι ε, θα μπορούσε να δοθεί λίγο πιο καλή κατεύθυνση, πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικός συμβιβασμό. Είναι σημαντικό να λέμε ότι υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία πίσω από την έκθεση αυτή που υποβάλλουμε. Όταν υπάρχει μια τέτοια εξεταστική επιτροπή είναι σημαντικό να υπάρχει ισχυρή υποστήριξη. Και τρίτον, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, δεν είναι αρκετό αυτό που κάνουμε, γιατί θα υπάρχουν νέα σκάνδαλα, νέα leaks, νέες αποκαλύψεις. Πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά μας. Ε, και συνεπώς υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας, ακόμη και αν τελειώσει στις 8 Δεκεμβρίου ε, η δική μας δουλειά και εκπνεύσει η εντολή μας, συνεχίζει η δουλειά μας. Εμείς ολοκληρώνουμε τη δουλειά μας, ε, όμως πρέπει να συνεχίσει μετά η δουλειά της εφαρμογής των πορισμάτων μας. Ευχαριστώ. Στο τέλος του σημείου 5 θέλω να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή, τους ε, συντονιστές, όλους τους και εισηγητές, αλλά κυρίως όλους τους συναδέλφους ε, που τους τελευταίους 18 μήνες συμμετείχαν. θα βγάλω και ένα κατάλογο παρουσίας από τη γραμματεία γιατί στην αρχή ο κόσμος ε, σκοτώθηκε να είναι μέλος στην Επιτροπή, αλλά στο τέλος η παρουσία δεν ήταν η ίδια. Να δούμε ποιες ήταν οι παρουσίες και στο μέλλον ε, ποια μέλη θα διορίζουμε σε αντίστοιχες επιτροπές. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, πάμε στο σημείο 6, διάφορα. Το λόγο έχει η Σάνφη Πατρίσια Σούλιν. Παρακαλώ. Eh, kratka se pa vezujem na vaše eh, uvodne besede, ko ste povedali da... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, πω δύο λόγια. Γιατί όσα ακούστηκαν μου θυμίζουν ότι σε μία από τις συνεδριάσεις του Οκτώβρη ναι, τα γερμανικά ακούγονταν. Ε, σε μία από τις συνεδριάσεις του Οκτώβρη είχε ανακοινωθεί ότι θα προχωρούσαμε στην εντοπισμό των ε, καταχρήσεων, από, κακοδιαχειρήσεων από το σλοβενικό τραπεζικό σύστημα. Να σας ενημερώσω ότι το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας ε, συνεδρίασε συνήλθε τον ε, Σεπτέμβριο και ετοίμασε, συνέταξε μια έκθεση για τον εντοπισμό ευθυνών στο σλοβενικό τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κάποιες λοιπόν ε, διευκρινήσεις. Η Νόφσκα Μπάνκα επέτρεψε σε έναν Βρετανό πολίτη Ιρανικής καταγωγής επί δύο χρόνια να στείλει χρήματα στο Ιράν, τη Ρωσία και άλλες τρίτες χώρες μέσω λογαριασμού του στη Σλοβενία. Τα χρήματα που προέρχονταν από τις χώρες αυτές έφτασαν στην Σλοβενία, στο λογαριασμό του στην Όβα Λιουμπλιάνσκα Μπάνκα και μετά μεταφέρθηκαν σε διαφορετικούς λογαριασμούς διαφόρων χωρών. Η τράπεζα αυτή, τράπεζα... Πρόεδρος, αποφασίσαμε στους συντονιστές να κάνουμε ακρόαση για το Αζερβαϊτζάν και ταυτόχρονα για τη Σλοβενία την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και σας παρακαλώ να μας δώσετε τα έγγραφά σας για να το προετοιμάσουμε. Και αφού τα εγκρίνει όλα αυτά η γραμματεία και τα, τα ελέγξει μάλλον, το πρωί στις 22 Νοεμβρίου ε, προγραμματίζουμε την ακρόαση. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν αίθουσες και διερμηνείς αλλά κανονικά 22 Νοεμβρίου, πριν λήξει η θητεία μας, θέλουμε να κάνουμε δημόσια ακρόαση για την περίπτωση της Σλοβενίας και του Αζερβαϊτζάν. Αυτό αποφάσισαν σήμερα το πρωί οι συντονιστές. Το είπα στην αρχή ε, σύντομα, χωρίς να αναφέρω ημερομηνία και θα σας ήμουν ευγνώμων αγαπητοί συνάδελφοι, να διαβιβάζετε τα έγγραφα Αυτό όχι μόνο στον Πρόεδρο και τη Γραμματεία αλλά και στους συντονιστές και στους εισηγητές. Εντάξει. Ε, vielen Dank, damit Ωραία. Νομίζω το μέλημά σα βρίσκει ανταπόκριση. Θα το συζητήσουμε σε δημόσια κρόαση. Vielen Dank, dann komme ε, ε- Ευχαριστώ πολύ. προσεχή συνεδριάσει. όπως είχαμε συμφωνήσει στην αρχή, αν πάνε όλα καλά και αν δεν διαφωνήσει κανεί μέχρι την Τρίτη, θέλουμε την Τετάρτη το απόγευμα 3 με 5,5 να εξετάσουμε και να ψηφίσουμε μάλλον τις τροπολογίες και τις συμβαστικές για να προετοιμάσουμε την, την έκθεση, να την ολοκληρώσουμε. Η έκθεση και τα παραρτήματα κατόπιν θα παραδοθούν στα χέρια των πολιτικών ομάδων. Θα έχουμε συζήτηση 23 του μηνός και συντονιστές και οι πολιτικές ομάδες πέρα από τις διαπιστώσεις έκθεσης θα πρέπει να κάνουν περαιτέρω πολιτικές συστάσεις όπως συμφωνήσαμε σήμερα το πρωί στους συντονιστές. Και η τελική μας συζήτηση θα γίνει στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ τη Γραμματεία και ιδιαίτερα τον κύριο Κόρβο που έχει ε, κάνει, ε, μάλλον έχει να καταρτήσει τις ε, λίστες ψηφοφορίας. Μέχρι αύριο θα πρέπει να τα έχει χτενίσει όλα αυτά. Πολύ δουλειά τον περιμένει. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, αλλά και τους δερμηνείς ο Πρόεδρος. Και κηρύσω επισήμως και το πέρας αυτής της συνεδρίας. Ευχαριστώ. εμείς ευχαριστούμε.